Και η επόμενη συνεδρίαση είναι αύριο 9 ε, Ιουνίου 2016, 9 ε, με 2 και 3 με 5. Ε, η μερίσια διάταξη έχει δημοσιευθεί και βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λήξης της συνεδρίασης. Καλό σας βράδυ και καλή σας νύχτα.